Όπως σας είπα νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης που μόλις ολοκληρώθηκε. Δυστυχώς χάσαμε προώρα το συνάδελφο Γιάννης Νίλσον. Σήμερα το πρωί απεβίωσε στη Σουηδία. Ύστερα από σύντομη ασθένεια. Ο κύριο Νίλσον πρωτοεκλέχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011, επανεξελέγει το 2014 και ανήκε στους κόλπους του Σουηδικού Σορδημοκρατικού κόμματος τη Σουηδίας και εδώ στου σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ήταν μέλος της επιτροπή των Μεταφορών, Περιφερειακών Υποθέσεων αλλά και της αντιπροσωπείας, για τη σχέση με τη Λευκορωσία. Ο κύριο Νίλσον ανέπτυξε την πολιτική του δραστηριότητα με γνήσιο ενθουσιασμό και μοναδική δυνατότητα ε, για ε, καταπώνηση και έργαση. Αγωνιζόταν για μια κοινωνική οικονομία, ένα ιδεώδες το οποίο πίστευε ακράδαντα. Που ήταν και ο αγώνας όλης του της ζωής. Στο όνομά σας θέλω να απευθύνω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τη σύζυγο και την κόρη του, τα θερμά συλληπιτήρια στους φίλους του, στους συντρόφους του, στην πολιτική του ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε όλους εκείνους που τον γνώρισαν, σε όλους εκείνους που τρέφουν που εκτίμηση στο πρόσωπό του και σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γέλς Νίλσον. Κυρία Ροντρίγκε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λαμβάνω το λόγο εκ μέρου τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ομάδα στην οποία ήταν μέλο ο κύριο Νίλσον. Πολύ λίγα λόγια. Θέλω καταρχά να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τιμή, για το λεπτό συγγύη. Θέλουμε εμείς, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, να τον θυμόμαστε όπως ήταν ένας άνθρωπος πολύ γενναιόδωρος, ένας άνθρωπος προσιλωμένος και στρατευμένος στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τρόπο να επικοινωνεί με τον κάθε άνθρωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνιζόταν για την κοινωνική οικονομία σε όλη την Ευρώπη. Το Γιάννη Νίλσον, πάντα έτσι θα σε θυμόμαστε θα σε θυμόμαστε πάντα με θερμά αισθήματα φιλίας. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Ο κύριος Φόξ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα σε όλους στην εκλογική μου περιφέρεια δολοφονήθηκαν με ένα ευρωπαραλυτικό ε, αέριο ένας άντρας και η κόρη του, αλλά και ένας αστυνομικός που έσπευσε στην περιοχή. Εχθές η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είναι πιθανόν να είναι υπέτεια για αυτήν την αποτρόπαια πράξη η Ρωσία, είτε απευθεία γιατί ε, παρήγγειλε μια τέτοια δολοφο... απόπειρα δολοφονίας ή ε, εξαμελίας διότι επέτρεψε να κυκλοφορεί αυτό το απαγορευμένο υλικό. Πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ρωσία και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και μια αφύπνιση για όλους μας. Δοκιμαζόμαστε εμείς στην Δύση, η προσάρτηση της ε, Κρυμαίας, κυβερνοεπιθέσεις στην Εστονία, η χρήση χημικών στο Σόλσπουρι δείχνουν ένα ανισχυτικό σχεδιάγραμμα δράσης το οποίο πρέπει να σταθούμε όλοι ενωμένοι και στεναροί. Ευχαριστώ. L'applauso della plenaria non ha bisogno di ulteriori commenti. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ε, κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε θέλω να αφαιρθώ στους κανόνες περί συμπεριφοράς των μελών του Κοινοβουλίου, που συμπεριφέρονται ένας εναντί του άλλου. Σήμερα το πρωί στη συζήτηση για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, ένα μέλος του Κοινοβουλίου, ο κ. Άλαν Σμιθ από τη Σκοτία, σωστά χρησιμοποίησε κάποια διατύπωση για να επικρίνει υπέρμαχους του Brexit όπως εγώ. Χρησιμοποίησε μια λέξη τη επικρίση του που θεωρώ ότι εσεί σαν πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου θα θεωρείτε ότι είναι πολύ ε, προσβλητική και ζητώ συγγνώμη. Είπε ότι ε, είναι... Είναι κάποιος ο οποίος ε, αποπατεί ουσιαστικά, αφοδεύει και και χρησιμοποιείται αυτό Σάιστερ για κάποιον που φοδεύει. Αλλά επίση έχει και κάποια εβραϊκή έννοια. Σάιστερ χρησιμοποίησε σαν λέξη. Επέκρινε τακτικά ε, του ε, Εβραίου. Του θεωρούσε ότι είναι ανηλικρινεί. Ήταν προσβλητική λέξη. σω δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη Σάιστερ ο κ. Σμιθ. Αλλά τώρα αναγνωρίζοντα τι ισχύ έχει αυτή η λέξη, θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη και πρέπει να το αναγνωρίσει ο ίδιο γιατί χρησιμοποιεί αυτή την προσβλητική λέξη. Κύριε Σμίθ, θέλετε να πείτε κάτι. Βέβαια, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ίσως να μην ξέρετε τη λέξη. Ποιο είναι ο ορισμό του Σάιστερ στο ε, λεξικό Κόλλιν. Σάιστερ ή Σάιστερ, πληθυντικό, αν αναφέρεστε σε κάποιον και του σε νομικό ή πολιτικό και τον πείτε Σάιστερ, εννοείται ότι είναι ανηλικρινή και ανήθικη κάποιος ειδικά δικηγόρος ή πολιτικός που ε, χρησιμοποιεί, ε, κινείται ανήθικα. Δεν αναφέρατε τίποτα για Εβραίους και δεν είχα κάτι τέτοιο υπόψη μου και αυτή η κατηγορία είναι γελία. Λοιπόν, την απορρίπτω αυτή την καταγγελία και παροτρύνω ε, το Σκηνοβούλιο να μην χρονοτριβεί πάνω σε αυτές τις ανοησίες. Ανήθικος δεν μπορεί να πει κανείς και ανήθικος. Δεν μπορεί να το πει κανεί σε κάποιον άλλον. Σε κανέναν δεν μπορεί να το πει αυτό σαν διατύπωση. Αν από την πλευρά σας δεν υπήρχε πρόθεση, καμία πρόθεση, ε, πιστεύω ότι τελικά η διευκρίνηση αυτή που έγινε είναι επαρκή, Ανήθικος και ανηλικρινής όμως ε, δεν μπορεί να απευθύνει ένα συνάδελφο στον άλλον σαν έκφραση. Ε, κύριε Ντάρτμουθ παρακαλώ. Κύριε Ντάρτμουθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε ε, το λόγο. Άρθρο 11, τμήμα 3. Λοιπόν, θα αναφερθώ στο άρθρο 11, 3. Και τι λέει ο εσωτερικό κανονισμό επ' αυτού. Ότι η συμπεριφορά των μελών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, λέει. Και ε, τώρα άκουσαμε τα σχόλια του κ. Σμιθ που ήταν επαρκή. Παρόλα αυτά, παραβίασε τις αξίες και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είχαμε εξαιρετικό παράδειγμα αυτού από τα σχόλια της ε, κυρίας Φόξ προηγουμένως, που τα τήρησε αυτά. Παρ' όλα αυτά ζητώ ο πρόεδρος, τον κύριο Σμιθ, ε, να τον ε, επιπλήξει επισήμως, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κύριε Μπόιλαν. Κυρία Μπόιλαν μάλλον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιμπραήμ Χελάουα που βρίσκεται στην εξώστη των καλεσμένων. Το Δεκέμβριο του 2015 ψηφίσαμε ένα ψήφισμα ζητώντα την άμεση απελευθέρωσή του και χαιρόμαστε ιδιαίτερω που είναι ελεύθερος πια, είναι εδώ μαζί μας σήμερα Σας ευχαριστούμε κυρία Μπόιλαν, ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Κόμπερν και μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Κόμπερν. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Συνήθως ε, δεν με ε, αναστατώνει τίποτα. Αλλά ο κύριος Σμιθ είναι πραγματικά ε, πολύ, είναι ε, πολύ επιδέξιος στα θέματα της πολιτικής ορθότητας και θα έπρεπε να προσέχει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι ξέφυγε, το παρατράβηξε και οφείλει στη συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι δεν περιπεί τιμή ούτε στον, ε, ίδιο, στον εαυτό του προσωπικό, ούτε στην πολιτική του ομάδα με τέτοια συμπεριφορά. Καλώς. Κύριε Κόμπεν, γνωρίζουμε ότι εσείς είσαστε αρκετά Ξέρουμε πώς ε, ε, δραστηριοποιείστε και ανάβετε. Εγώ θα ήθελα να θέσουμε τέρμα σε αυτό. Ξέρω ότι η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος ε, ήταν από πολιτική σκοπιά και δεν είχε σκοπό να προσβάλλει τον συνάδελφο. Από την ερμηνεία που άκουσε πρόκειται, πρόκειται περί πολιτικής επίκρισης και δεν ήθελε να προσβάλλει ούτε για λόγους ρατσιστικούς, ούτε για λόγους πολιτικούς δεν ήθελε να προσβάλλει. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ερμηνευτεί η λέξη αυτή σαν ε, πολιτική επίκριση. Αν ήταν διαφορετικά θα πρέπει να παρέμβουμε. Πιστεύω ότι πρόκειται ε, περί ε, κρίσεως πολιτικής, κρίσεως πολιτικής και δεν ήταν τίποτα περισσότερο. Και τώρα πάμε στην ψηφοφορία.